Καλημέρα σε όλες τις γλώσσες από την Πρόεδρο. Έλα. Κυρία Ταραμπέλα, θα αρχίσουμε. Καθίστε παρακαλώ. Πρώτα απ' όλα, Έχουμε μία πρόταση αλλαγή ε, ημερήσια διάταξη ε, διάταξης. Αποφασίσαμε χθε στους συντονιστέ. Θα προσθέσουμε δύο τροπολογίες της κυρίας Βένσον για το σχέδιο έκθεσης Επιτροπής ΙΜΚΟ για την ε, κοινή αγορά για τους Ευρωπαίους. 7 Φεβρουαρίου είναι η προθεσμία για την Επιτροπή ΙΜΚΟ. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχουμε για να ε, επηρεάσουμε τις εξελίξεις στην Επιτροπή ΙΜΚΟ για αυτή την έκθεση. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, θα το προσθέσουμε αυτό το σημείο μετά το 12, γιατί είχε κυρωθεί χθε το 13, θα είναι το σημείο λοιπόν 12α. Αρχίζουμε την ε, ψηφοφορία. Ελπίζω να έχετε φέρει και τις κάρτες σας μαζί. Σημείο 8. Ε, ε, Το πρώτο σημείο είναι το 13, διορθώνει η Πρόεδρος, ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση 2010. Η συγκεκριά μας είναι η κυρία Νενταλτσέβα Παρακαλώ, κυρία μου, αν θέλετε το λόγο. No. Όχι, όχι. Ας ε, περάσουμε ευθύς αμέσως στην ψηφοφορία. Είστε έτοιμοι. E Για να διευκολύνω την ψηφοφορία, γιατί έχουμε και μπόλικες, ε, θα αναφέρομαι μόνο στον αριθμό της τροπολογίας. Υπαριθμό 47, παρακαλώ. Ποιοι είναι υπέρ? Κατά. ηλεκτρονική ψηφοφορία για να κάνουμε μια επαλήθευση. Παρακαλώ. Against? Votes is random. Ε, πέραση ψηφοφορίας. Απερίφθη. Θα ήθελα να ε, ψηφίζετε με μεγαλύτερη σαφήνεια αν θέλετε, να φαίνεται τι ψηφίζετε για να διευκολύνουμε τις ψηφοφορίες. Ε, τραπολογία 48 υπέρ παρακαλώ. Κατά Αποχές. Εγκρίθηκε. Ε, της Επιτροπής η 1. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Η 4 της ίδιας Επιτροπής. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται επίσης. Η παριθμόν 8. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίθηκε η 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 50 υπέρ Η 49 διορθώνει πρόεδρος της κυρίας Παρβάνοβα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 50. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. η 2 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η 51. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 11 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά Θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Παρακαλώ ξαναψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Η 12 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 20 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ. Πέρα, εγκρίνεται. Η 52 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά θα κάνουμε την επαλήθευση, παρακαλώ, για την 53. 53. Για την 53. Πέρας. Απερίφθη τελικά. Η 54 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. επαλήθευση, ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. Η 19 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 55 υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται, η 30 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 33 της απασχόλησης υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, η 56 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, η 57 υπέρ, κατά, Αποχές απορρίπτεται 58. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 18 της απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 28 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 59 υπέρ Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 60 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 62 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 14 Επιτροπής Απασχόληση υπέρ. Κατά. Αποχές θα κάνουμε την ηλεκτρονική επαλήθευση, παρακαλώ, για τη 14 της Επιτροπής Απασχόλησης. 14, έτσι. Κατά. Θα επαναλάβουμε την ψηφοφορία για την 14 της επιτροπή Απασχόλησης, παρακαλώ. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 25 υπέρ. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 65 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 66 και η 27 της Επιτροπής Αποσχόλησης ταυτόσημες υπέρ κατά αποχές θα κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Για την 66 και την 27 της Επιτροπής Αποσχόλης Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίθηκαν. 67 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 68 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Η 7 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 17 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ, κατά αποχές επαλήθευση, επαλήθευση. Για τη 17 της Επιτροπής Απασχόλησης. πέρες ψηφοφορίας. Εγκρίθηκε. 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. εβδομήντα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. 71. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 3 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές επαλήθευση Νομίζουμε ότι απορρίπτεται, αλλά ας επαληθεύσουμε. Πέρας ψηφοφορίας. Όντως, όντως. Γιατί συνάδελφος από τους φιλελεύθερους καταψήφισε την ε, τροπολογία 74 υπέρ κατά Αποχές εγκρίνεται. 31 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι απορρίπτεται επαλήθευση. Παρακαλώ για την 31 της Επιτροπής Απασχόλησης. Πέρας. Απορρίπτεται. 21 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ κατά επαλήθευση παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ Ah. Εγκρίνεται ε, με την ψήφο της κυρίας Νικολάη. Ήταν υπέρ, υπέρ, υπερψηφίσατε την τροπολογία, έτσι δεν είναι. Ωραία. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 22 της Επιτροπής Αποσχόλησης, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 78 υπέρ. 78. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμφιβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα 82, η 82 υπέρ. 82 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 84 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 86 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 34 Επιτροπής Απασχόλησης. ό,τι δεν χρειάζεται να ψηφίσουμε. 88 υπέρ. Κατά. Αποχές Απορρίπτεται 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 87 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 της Επιτροπής Απασχόλησης. Σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα δεν θα το ψηφίσουμε γιατί καλύπτει την τροπολογία 87-91 τροιπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία για επαλήθευση, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Είναι 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 35 35 σε δύο τμήματα, το πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται γι' αυτό, 93 υπέρ, κατά, φιλελεύθεροι. Είναι 93 ψηφίζουμε. Υπέρ. Υπέρ εγκρίνεται λοιπόν. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 95 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 29 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές επαλήθευση παρακαλώ άρχεται ψηφοφορία για την 29 πέρας απερίφθη 23 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 15 το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 υπέρ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 101 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 106 υπέρ. Και ή την 107 μαζί. Όχι χωριστά. Μόνο την 106 παρακαλώ. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 109 υπέρ κατά κατά αποχές εγκρίνεται 110 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 111 ματέρα υπέρ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 112 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 113 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 114 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 115 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 36 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 η 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 26 της Επιτροπής απασχόληση δεν θα την ψηφίσουμε στην 24 πάμε 24 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 25 με προφορική τροπολογία ε, υπάρχει η ένσταση για την προφορική τροπολογία. Είναι κάποιο κατά. Όχι. Ωραία. Με την προφορική τροπολογία ψηφίστε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 26 σε δύο τμήματα. Το πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και τώρα η 34 Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 35 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 36 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 37 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 40 καταπίπτει. Ζητήθηκε επαλήθευση ηλεκτρονική για την 41. Παρακαλώ ψηφίστε. Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. 40, 40. Euh, euh, υπέρ. Κατά. Αποχή συγκρίνεται. 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 44 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 43 σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 46 σε δύο τμήματα το πρώτο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρώτη τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τέσσερα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Πέντε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 Την 11 ψηφίσαμε μόλις τώρα. Αν θέλετε ομού να τις ψηφίσουμε τις τροπολογίες από την 12 έως και την 17. Συμφωνείτε? Υπέρ όλων αυτών των τροπολογιών. Λοιπόν, διόρθωση της Προέδρου από τη 12 έως την 15 ομού. Ψηφίστε παρακαλώ. 12, 13, 14, 15. Υπέρ. 12, 13, 14. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Η 15 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ορίστε. 16 και 17 μαζί υπέρ. Κατά. Μόνο για τη 16 υπέρ κατά, αποχές, εγκρίνεται, 17, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται και αυτή. Ε, θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά τώρα για την τελική ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται με 22 ψήφους υπέρ 2 κατά και καμία αποχή. Συγχαρητήρια, κυρία Νεντελσέβα. Και τώρα Τώρα θα περάσουμε στο σημείο 8. Απαλλαγή 2009. Γενικό προπολογισμό τη ΕΕ, ε, τμήμα 3, Επιτροπή. Η κυρία Ιράτσε Γκαρσία Πέρες είναι η συγγήτριά μας. Θα ψηφίσουμε. Προτείνω όμου να ψηφίσουμε μέχρι την παράγραφο 5. Υπάρχουν αντιρρήσεις. Ας ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η παράγραφος 5 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία, τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Ε, εγκρίνεται με 24 ψήφους υπέρ, 0 κατά, 0 αποχές. Συγχαρητήρια κυρία Πέρες. Και τώρα στο επόμενο σημείο το 9... και έκθεση 2010 σχετικά με την υλοποίηση των προγραμμάτων της πολιτικής για τη συνοχή 2007 ως 2013. Ε, δεν παρίσταται ο γιατί Θα περάσουμε απευθεία στην ψηφοφορία. Τροπολογία 1. Α, μπορούμε όμως να ψηφίσουμε πάρα πολύ ωραία. Πέντε τροπολογίες είναι. 1, 2, 3, 4, 5. Ναι, υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνονται. Και δεν χρειάζεται τελική ψηφοφορία γιατί είναι μόνο οι τροπολογίες. Τώρα, σημείο 10. Η εξωτερική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής προώθηση του εργατικού δικαίου, δικαίου συγγνώμη, των κοινωνικών προτύπων και ε, η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων. Μόνο τις τροπολογίες και πάλι θα εγκρίνουμε εδώ. Δεν υπάρχει τελική ψηφοφορία. Ας ψηφίσουμε ομού επίσης Τέσσερις τροπολογίες υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνονται. Σημείο 11. Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή απασχόληση. Κυρία Παπαδοπούλου, θέλει το λόγο, είναι η συγγετριά μας. Θέλετε το λόγο? Παρακαλώ. Έχουμε υποβάλει αυτό το σχέδιο γνωμοδότησης. Η τροπολογίες η αρμόδια επιτροπή επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Ελευθεριών Πολιτικών Δικαιωμάτων κλπ. Οι περισσότερες τροπολογίες τις οποίες έχω μελετήσει είναι αποδεκτές εκτός από μερικές ε, τις οποίες διαφωνήσαμε ως ομάδα σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, τροπολογία 7 ζητάει την αποφυγή των διακρίσεων για εποχιακούς εργάτες σε αντίθεση με εργάτες που εργάζονται σε άλλους τομείς και για την τροπολογία 19 υπάρχει προφορική τροπολογία για την διαγραφή μέρους της παραγράφου. 7, 19 και αν προσέξετε υπάρχει στη 19 μία διαγραφή η οποία λέει που θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μέχρι ότου τιμωρηθούν punished. Εκεί όλη αυτή η πρόταση διαγράφεται. Αυτή είναι η πρόταση δηλαδή. Και υπάρχουν άλλα σχόλια για τροπολογίες το 26, 17, 20 και δεν, δεν τις έχω δεχθεί για διαφορετικούς λόγους. 26 την απορρίπτω, διότι η ελευθερία ε, ε, πρέπει να διατηρηθεί, το Freedom of Association, το 17 επίσης απορρίπτεται, διότι προτιμώ το κείμενο της Κομισιόν, διότι υπεραμείνεται μια ομοιόμορφης προσέγγισης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το 17 επίσης εισάγει την αρχή της επικουρικότητος και στο 20 και στο 18, τροπολογίες 18 και 20 επίσης τις απορρίπτω. Δεν συμφωνώ με το περιεχόμενό τους. Γιατί λέει ότι οι αλλοδαποί, οι τρίτων χωρών ε, θα πρέπει να μπορούν να παραμείνουν έστω και με διαφορετικές μορφές θεωρήσεων. Αυτό αντιτίθεται στη γενική έννοια ε, της ε, προτάσεως. Είμαστε λοιπόν κατά των εξαιρέσεων και γι' αυτό απορρίπτω και το 20. 26, 17, 18, 20 δεν τις ε, Οι σοσιαλιστές είναι υπέρ. Περνάμε στην ψηφοφορία παρακαλώ. Η 7 απεσύρθη έτσι οπότε 8 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 9 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται επίσης 24 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται η 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 25 ε, καταπίπτει 26 κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 14 υπέρ. 27 καταπίπτει, γι' αυτό δεν την ανέφερα. 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 15 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Η πρώτη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η δύο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η τρία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά κατά αποχές απορρίπτεται. 18 υπέρ Κατά. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 19. Με προφορική τροπολογία είναι 19. Αν δεν υπάρχουν ενστάσεις, παρουσιάστηκε ήδη η προφορική τροπολογία, θα ψηφίσουμε υπέρ. Κατά. Κατά παρακαλώ. Αποχές εγκρίνεται. Η τέσσερα. Υπέρ. Επίσης με προφορική τροπολογία η τέσσερα. αν δεν υπάρχουν αστάσεις. Ας ψηφίσουμε με την προφορική τροπολογία για την τέσσερα. έτσι υπέρ. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η είκοσι υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, η 5 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 21 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 22 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, 6 υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Η 23 ψήφοι υπέρ, καμία κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Παπαδοπούλου. Euh, Ευρωπαϊκή συνεργασία τώρα στο επόμενο σημείο στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση για την υποστήριξη στρατηγική Ευρώπη 2020. Η κυρία Σένισιν είναι η συγγήτριά μα. Δεν θέλετε το λόγο. Όχι. Ευχαριστούμε και περνάμε κατευθείαν στην ε, ψηφοφορία. δεν Μπορούμε να ψηφίσουμε ομού την πρώτη σελίδα των τροπολογιών στη λίστα της ψηφοφορίας. Την τρίτη και την τέταρτη εννοείται, λέει η Πρόεδρος. Vamos então votar 4. Την τέσσερα Υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ, πέρας. Εγκρίθηκε. Η τρία υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Η πέντε υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται. Τώρα 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12 ομού ψηφίστε. Όχι, 6, 7 και 9 μόνο. Υπέρ.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 Επαλήθευση παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 28. 28 καταπίπτει. Και 27. Και 26. 29 τότε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται η 1. Υπέρ. Κατά απόχες εγκρίνεται 2 υπέρ κατά απόχες εγκρίνεται επίσης τελική ηλεκτρονική ψηφοφορία τώρα παρακαλώ ψηφίστε παρακαλώ πέρας 23 είναι η ψήφοι υπέρ, καμία κατά, καμία αποχή. Συγχαρητήρια κυρία Σένιτσεν.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 για το σημείο 12α, έτσι, την αλλαγή που κάναμε στην ημερήσια διάταξη στην αρχή της συνεδρίασης για την ενιαία αγορά για τους Ευρωπαίους. Είναι δύο τροπολογίες ε, της κυρίας Βένσον. Μπορούμε να ψηφίσουμε σας παρακαλώ. Είστε έτοιμοι. Μαζί θα τις ψηφίσουμε και τις δύο τροπολογίες υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνονται και οι δύο. Τώρα, στο 13 θα περάσουμε τώρα, έτσι δεν είναι. Το 13 το έχουμε ήδη κάνει. Το 14. Το πρόσωπο της γυναικείας φτώχεια στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η κυρία Πλάμ είναι η συγγήτριά μας. Θέλετε το λόγο, παρακαλώ. Thank you, Chair. <clears throat> I would... Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ καταρχάς όλους τους συναδέλφους για τη στενή του συνεργασία σε αυτή την έκθεση. Είναι μια σημαντική έκθεση και ευχαριστώ και τη Γραμματεία της Επιτροπής. Θεωρώ ότι εάν υιοθετήσουμε αυτή την έκθεση θα έχουμε προχωρήσει ένα βήμα για να εφαρμόσουμε, να υλοποιήσουμε την ισότητα των φίλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή λοιπόν αντιπροσωπεύει ένα βήμα πρόοδου, σας ζητώ να την υπερψηφίσετε γιατί προτείνει πολλές λύσεις για την επίτευξη αυτού του σημαντικού στόχου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Περνάμε στην ψηφοφορία. Η 39. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 40 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 1 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 42 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 3 της Επιτροπής Απασχόληση υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 9 της Επιτροπής Απασχόληση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 33 της Επιτροπής αποσχόληση υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 44 τώρα 44. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. Η 46 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές Επαλήθευση παρακαλώ. Ψηφίστε παρακαλώ. Για τη 46 ψηφίζουμε. Ταυσάδα από Πέρας ψηφοφορίας. Τρεις υπέρ, τρεις κατά και 17 αποχές με την ισοψηφία απορρίπτεται. Η συμβαστική 2 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα, στην 50 δεν πάμε. 50 υπέρ. Κατά, αποχές εγκρίνεται. 51 υπέρ. Κατά, αποχές επαλήθευση. Επαλήθευση ηλεκτρονική. Πέρας. Foi e Εγκρίθηκε. 52 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 54 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται.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 Συγγνώμη, δεν κοιτάτε καθόλου μέσα στην αίθουσα. Κάντε τη μόνη σα την ψηφοφορία. Μα είναι τρει τελευταίε ψηφοφορίε, ούτε καν κοιτάτε τι, γίνεται μέσα στην αίθουσα. We voted uh, the compromise. Τη συμβαστική 15 τώρα ψηφίζαμε, αλλά δυστυχώ τα υπόλοιπα σχόλια είναι εκτό μικροφώνου. Δεν τα ακούμε εμεί. Ε, Θα ψηφίσουμε και πάλι για τη συμβαστική 15. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 60. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 61. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Επαλήθευση θέλετε. Ορίστε. Για την 61. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέραση encerrada a Πέρας ψηφοφορίας. Rejeitado. Απορρίπτεται. Η ψηφία απορρίπτεται. 141 ε, τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 142 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 146 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 62 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Η συμβαστική 3 τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τώρα 63 παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Επόμενη σελίδα παρακαλώ. Η 66. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 67 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αλλά ας το επαληθεύσουμε καλύτερα. Αρχίστε παρακαλώ, ψηφίστε παρακαλώ, πέρας ψηφοφορίας. Επρουβάδα. Ναι, όντω εγκρίθηκε. 68 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η 10 της επιτροπη απασχόληση υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 34 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 71 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η 69 υπέρ. Κατά. Αποχές. Κρίθηκε. Ε, καλά, ζητείτε επαλήθευση. Για την 69 ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. Η 70 τώρα. Υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται 72 υπέρ. Όχι, 72 καταπίπτει, 73 υπέρ. 73 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές, Άλλοι πώς ψηφίσατε φιλελεύθεροι υπέρ, υπέρ, ε, εγκρίθηκε, 75 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 76 υπέρ. Κατά αποχές ε, εγκρίνεται 77, 78 και 79 είναι τρεις ταυτόσιμες τροπολογίες. Ψηφίστε εκεί για τις τρεις υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Θα κάνουμε την επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Ναι, ναι, εγκρίθηκαν. 80. Η 80... Όχι, καταπίπτει. Κατέπεσε. Η 82. 82 τώρα. Της κυρίας Γκαρσία Πέρες. Υπέρ. Κατά. Αποχές, επαλήθευση παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, εγκρίθηκε. 83 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 4 υπέρ, κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Γιατί είναι και συμβαστική τροπολογία. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονική, παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 84. Είναι προστίκη. 84. Υπέρ παρακαλώ. 84. Τροπολογία 84. Αμέσως μετά τη συμβαστική 4. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση, ε, ηλεκτρονική επαλήθευση σας παρακαλώ. Πέρας. Α, περίφθη. 88 τώρα. Της κυρίας Ματέρα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Είσαι 145 της κυρίας Γκαρσία Πέρες υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα. Η 90 στην επόμενη σελίδα. 90 της κυρίας Νικολάη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 14. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η, της Επιτροπής Απασχόλησης είναι τώρα όχι 91 ως προσθήκη 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται η 7 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε η, ε, της Επιτροπής Απασχόλησης 11 τώρα ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Η 36 της ίδιας επιτροπής υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Η συμβαστική 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην επόμενη σελίδα περάστε παρακαλώ. Η τροπολογία 104 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 καταπίπτει. Η 105 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 106 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ηλεκτρονική άρχεται ψηφοφορία ε, για την 107 έτσι τα Πέρας ψηφοφορίας. Απερίφθη. Η 8 της Επιτροπής Απασχόλησης. Α, δεν θα την ψηφίσουμε. Συμβαστική 6. 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Επόμενη σελίδα παρακαλώ. Η 15 της Επιτροπής Απασχόλησης υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 112 καταπίπτει. 113 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση παρακαλώ για την 114. Παρακαλώ. Πέρας. Απορρίπτεται. 12 υπέρ, 12 κατά, ψηφία, απορρίπτεται. 115 τώρα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 121 σκυριάς πλάμ ε, ε, υπέρ κατά Αποχές. Εγκρίνεται. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 125 καταπίπτει. 126 τρώει υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 127 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 128 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 129 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 133 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επαλήθευση Ψηφίστε ηλεκτρονικά παρακαλώ για την 133 για να γίνει επαλήθευση. 133. Πέρας. Εγκρίθηκε. Οι 134 και 35 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίστε για τις δύο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτονται και δύο. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Νομίζω ότι εγκρίθηκε επαλήθευση για την 136. πέρασε. Εγκρίθηκε. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Άποχες εγκρίνεται. Η 140 τώρα το πρώτο κομμάτι. Πρώτο τμήμα, συγγνώμη. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η 89 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 143 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 147 ε, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η πρώτη τροπολογία της κυρίας Γκαρσία Πέρες ε, με μια προφορική τροπολογία. Ε, ψηφίστε παρακαλώ υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Η τρία τώρα. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η δύο καταπίπτει. Η τέσσερα επίσης. Η πέντε τώρα. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Επαλήθευση. Ψηφίστε παρακαλώ. Alteração 5. Η 5 πέρας. Εγκρίθηκε. Η 8 υπέρ. Κατά απόχες απορρίπτεται η 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 6 καταπίπτει η 10 τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 14 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 20 υπέρ κατά κατά παρακαλώ Επαλήθευση για την 20 παρακαλώ ψηφίστε Está encerrada a votação. Peras. Foi adotado. 19. Εγκρίθηκε 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 11. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η συμβαστική 12. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καλά, υπαλήθευση. Για την 25. Για την 25 παρακαλώ. Πέρας. Εγκρίθηκε. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 26. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Καταπίπτει 29 της Επιτροπής Απασχόλησης, όχι δεν την ψηφίζουμε. 31 τώρα, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 33 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση ψηφίστε παρακαλώ πέρας να, απερίφθη η 13 τώρα σημαστική υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τελική ψηφοφορία παρακαλώ ηλεκτρονική ψηφοφορία άρχεται πέρας 23 ψήφοι υπέρ, μία κατά. Συγχαρητήρια στην κυρία Πλάμ. Τώρα, αυτό αναβλήθηκε για την επόμενη συνεδρίαση. Ένα λεπτά πριν τελειώσουμε. Θα ήθελα να σας θυμίσω και πάλι ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει τη 31η Ιανουαρίου, τη Δευτέρα, από τις 3 ως τις 6.30. Μια ακρόαση είναι για την κατάσταση των μητέρων που μεγαλώνουν μόνο τα παιδιά τους. Την 5η στις 3 Μαρτίου, την 5η, όπως έλεγα, από τις 9 ως τις 12.30 είναι ε, ο εορτασμός της Παγκόσμιας ημέρας της γυναίκας. Και για φέτος το θέμα είναι οι γυναίκες στην πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κ. Μπούζεκ, θα κάνει αρκτήρια δήλωση και η Μέρι Ρόμπινσον θα ε, παρευρεθεί πρώην ε, ε, πρωθυπουργός της Ιρλανδίας, θα είναι η βασική ομιλήτρια θα λάβετε και γραπτές ε, ε, πληροφορίες για την ακρόαση. Λύεται η συνεδρίαση μετά από αυτό και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.